Είναι πολύ σημαντική η ψηφοφορία που θα λάβει η χώρα τόσο λίγο. Αγαπητοί συνάδελφοι, εντό ολίγου θα αρχίσει η ψηφοφορία μας. Σας παρακαλώ θερμά καθίστε στις θέσεις σας. Συνάδελφοι, τέρμα οι συζητήσεις και καθίστε παρακαλώ στις θέσεις σας. Επανάληψη των εργασιών. Έναρξη της ψηφοφορίας. Η μερίσια διάταξη προβλέπει την ψηφοφορία επί της Συμφωνίας Πλαίσιο για τη σχέση μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής. Για την επόμενη κοινοβουλευτική θητεία. Θα ήθελα να ψηφίσουμε το κοινό ψήφισμα. Ποιος είναι υπέρ του ψηφίσματος για τη Συμφωνία Πλαίσιο. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Σας ευχαριστώ. Εγκρίνεται το ψήφισμα. Και τώρα θα ζητούσα από τον ε, πρόεδρο Θα ζητούσα από τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τον κύριο Ζωζέ Μανουέλ Μπαρόζο ε, να λάβει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πριν από λίγους μήνες ε, ε, στο πρόγραμμά μου που παρουσίασε εδώ στην Ολομέλεια πρότεινα να υπάρξει ειδική συνεργασία ανάμεσα στο Κοινοβούλιο και την Κομισιόν σε ένα νέο επίπεδο και πρότεινα τότε να ενισχυθούν περαιτέρω οι σχέσεις μας με θετικό τρόπο έτσι ώστε να αντικατοπτρίζουν τη νέα συνθήκη και το νέο αίσθημα που έχουμε ε, για τη διαμόρφωση της Ευρώπης. Τις τελευταίες εβδομάδες είχα σε βάθος συζητήσεις με μια ομάδα διαπραγματευτών των οποίων ηγήθηκε κύριο Λένα που ορίσατε εσείς για την αναθεώρηση τη συμφωνίας πλαίσιο. Αντράτω λοιπόν την ευκαιρία για να ευχαριστήσω όλους αυτούς ε, για τι ουσιαστικέ συζητήσει, αλλά και για την επικοδομητική του προσέγγιση. Είμαι βαθύτατα ικανοποιημένο, για το ότι πλέον βρήκαμε ε, συμφωνία ε, για τι αρχέ που θα διέπουν το έργο μα κατά τα επόμενα έτη. Θα ενισχυθεί η συνεργασία μας, σεβόμενη πλήρως τη θεσμική ισορροπία που διασφαλίζουν οι διασφαλίζει η συνθήκη. Ω πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εγώ προσυπογράφω τι αρχέ που αναφέρονται στην, ε, στο ψήφισμα που μόλι εγκρίνεται. αυτέ θα με κατευθύνουν, κυρίω όσον αφορά ε, την αναθεώρηση τη νέα συμφωνία πλαίσιο. Με την ε, έγκριση αυτού του ψηφίσματο με τόσο εντυπωσιακή πλειοψηφία, είμαι ακράδαντα πεπισμένο ότι έχουμε πλέον μια ικανοποιητική βάση για να ενισχύσουμε τι σχέσει μα. Για τα θέματα που αφορούν όχι μόνο του δύο θεσμού αλλά και το Συμβούλιο, Ειλικρινά ελπίζω ότι το Συμβούλιο θα προσχωρήσει και αυτό στην κοινή μας προσπάθεια για να βελτιωθεί το έργο όλων των θεσμών προς όφελος του συνόλου της Ευρώπης. Αν αργότερα σήμερα εγκρίνεται το νέο σώμα των Επιτρόπων, ε, θα ζητήσω από τον κύριο Σεύκοβιτς να ηγηθεί των διαπραγματεύσεων εξ ονόματος Επιτροπής για την αναθεώρηση της Συμφωνίας Πλαίσιο. Και επιθυμώ να σας διαβεβαιώσω ότι είναι εξίσου προσιλωμένος όπως και εγώ ε, και όλο το σύνολο των Επιτρόπων επιθυμεί να υπάρχουν αποτελεσματικές διαπραγματεύσεις. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ήταν πολύ θετική η προσέγγιση σας για τις διαπραγματεύσεις και θα ήθελα εκ μέρους ε, όλου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να, ευχαριστήσω θερμά την διαπραγματευτική μας ομάδα με επικεφαλή τον κύριο Λένε. Σας ευχαριστώ θερμά αγαπητοί συνάδελφοι όλους όσους τόσο θερμά κατά στις διαπραγματεύσεις. Συνάδελφοι, δεν έχουμε ακόμη νομοθετική πρωτοβουλία με βάση τη συνθήκη της Λισαβόνας. Αλλά ακούσαμε τις υποσχέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, που ικανοποιεί και τις δικές μας ε, φιλοδοξίες και έχουμε πια τη δέσμευση όχι μόνο του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά και των Επιτρόπων και πρόσκληση του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και το Σώμα των Επιτρόπων και το θέμα της ε, κοινή μας συνεργασίας με τα Εθνικά Κοινοβούλια. Και είναι πολύ σημαντικό γιατί η αρχή της επικουρικότητας είναι προσφυλή σε όλους μας. Χρειαζόμαστε και μελέτη επιπτώσεων για να βελτιώσουμε τη λειτουργία μας όπου δει και από αυτή την άποψη πιστεύω ότι θα ενισχυθούμε και θα προχωρήσουμε τη συμφωνία μας. Πάντως η συμφωνία αυτή δημιουργεί βάσιμες ελπίδες σε όλους μας ότι θα κάνουμε ό,τι μπορούμε και ό,τι χρειάζονται οι πολίτες μας για το μέλλον. Διακοπή τώρα μέχρι τη μιάμιση για τις υπόλοιπες ψηφοφορίες. Σας ευχαριστώ.